Ε, ε, ο εισηγητής είναι όντως ο κύριος Φερέιρα, όπως προανέφερα, όμως ε, δεν δύναται να παρευρεθεί και γι' αυτό ο κύριος Σιλικιώτης θα πάρει το λόγο. Ε, αγαπητοί συνάδελφοι, δυστυχώ ο εισηγητή τη έκθεση, ο συνάδελφο Ζωάου Φερέιρα, δεν μπόρεσε να είναι σήμερα μαζί μα. Γι' αυτό θα παρουσιάσω εκ μέρου του του κύριου στόχου που προωθούνται μέσα από αυτήν την έκθεση. Να επισημάνουμε αρχικά πω η έκθεση λαμβάνει υπόψη την έκθεση τη Κομισιόν με τίτλο καινοτομίο στα πλαίσια της γαλάζιας οικονομίας αξιοποίηση του δυναμικού των θαλασσών και των ωκεανών μας με στόχο την πρόθεση της απασχόλησης και της μεγέθυνσης ένα έγγραφο που έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης αφού έχει περιορισμένο πεδίο εφαρμογής και δεν καλύπτει όλους τους τομείς. προστίθενται λοιπόν τα πιο κάτω καινούργια στοιχεία. εκφράζεται δυσαρέσκεια για το βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο αντίκτυπο που θα έχουν στα εθνικά προγράμματα έρευνας οι περικοπέ των δημόσιων επενδύσεων στον τομέα της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας. ζητείτε τα αποτελέσματα της έρευνας που χρηματοδοτείται με δημόσια κονδύλια να αποτελούν δημόσια ιδιοκτησία για μη εμπορικού σκοπού και η αρχή αυτή να είναι δεσμευτική για τους εταίρους στα ερευνητικά προγράμματα τη ένωση. απορρίπτονται οι περικοπέ στον προπολογισμό του προγράμματο πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία του ορίζοντα 2020, τις οποίες τι οποίε πρότεινε η επιτροπή. η ορθή ανάπτυξη τη γαλάζια οικονομία απαιτεί αξιοπρεπή επαγγέλματα που συνδέονται με αυτήν και τη δημιουργία ποιοτική εργασία με δικαιώματα. στην έκθεση λοιπόν παροτρύνεται η κομισιόν και τα κράτη μέλη να εσωματώσουν τη διάσταση του φύλου σε όλα τα στάδια ανάπτυξη τη γαλάζια οικονομία καθώ και να και την πραγματική συμμετοχή των γυναικών σε αυτήν καλείται η επιτροπή να προσδιορίσει όλα τα ευρωπαϊκά κονδύλια που διατίθενται για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της γαλάζιας οικονομίας και να τα συγκεντρώσει σε μια ενιαία πλατφόρμα στην οποία θα έχουν πρόσβαση όλοι οι πολίτες. επίσης τονίζεται ότι η κομισιόν πρέπει να προβλέψει κονδύλια για καινοτομία και γαλάζια ανάπτυξη με σκοπό να χρηματοδοτηθούν η βασική έρευνα η επαγγελματική κατάρτιση η δημιουργία θέσεων εργασίας οι νεοσύστατες επιχειρήσεις οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας οι συνεταιρισμοί η εκπαίδευση η μείωση της φτώχειας των παράκτιων ζωνών η ανάπτυξη της βιοτεχνολογίας οι μεταφορικές συνδέσεις η ενεργειακή διασύνδεση η παράκτια πρόσβαση σε ευρυζωνικές υπηρεσίες η προστασία του περιβάλλοντος και η εμπορική εκμετάλλευση των καινοτόμων προϊόντων υπηρεσιών και συνεργασιών. αγαπητοί συνάδελφοι οι επενδύσει στην γαλάζια οικονομία θα πρέπει να επικεντρωθούν μεταξύ άλλων στην οικολογική καινοτομία στην αποδοτικότητα της χρήσης πόρων την κυκλική οικονομία τη διατήρηση της φύσης την προστασία του θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτή και τη βιώσιμη χρήση των πόρων. Στην έκθεση λοιπόν ζητείται από την Επιτροπή να ενσωματώσει τις αρχές αυτές στα εφιστάμενα καθώς και στα μελλοντικά προγράμματα στήριξη. εξίσου σημαντικό είναι το να καταρτιστεί κατάλληλο χρηματοδοτικό πλαίσιο προκειμένου να τονωθεί η καινοτομία η αφόρος ανάπτυξη της γαλάζιας οικονομίας και η δημιουργία απασχόλησης. το πλαίσιο αυτό θα συνδυάζει θα συντονίζει και θα διευκολύνει την πρόσβαση στα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία δημόσια ιδρύματα τοπικές αρχές αλλά και επιχειρήσει ιδίω μικρομεσαίες επιχειρήσει μη κυβερνητικέ οργανώσεις, για να υπάρξει έτσι ευρεία ενημέρωση για τις υφιστάμενες ευκαιρίες. είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε πως οι δημόσιες επενδύσεις διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην πρόθεση της ανάπτυξης και την πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού της γαλάζιας οικονομίας. πρέπει λοιπόν να ενισχυθούν χωρίς αυτό να σημαίνει πως θα παραγνωρίσουμε τον ρόλο των ιδιωτικών επενδύσεων πολύ σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν επίση οι δημόσιε εταιρείε ή οι εταιρείε που ανήκουν κατά πλειοψηφία στο κράτο σε τομεί όπω η εμπορική ναυτιλία η διαχείριση των λιμένων η ναυπηγική και τα έργα θαλάσσια και παράκτεια προστασία. απορρίπτουμε λοιπόν την εστίαση μόνο στον ιδιωτικό τομέα. όλα αυτά τα σημεία συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση και γι' αυτό καλούμε του συναδέλφου να την υπερψηφίσουν ώστε να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή πολιτική για τη γαλάζια οικονομία. ευχαριστώ πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Μαριάς για ένα λεπτό παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, η έκθεση πραγματικά είναι ενδιαφέρουσα και θίγει πάρα πολύ σημαντικά σημεία. Η γαλάζια οικονομία καλύπτει ένα ιδιαίτερο ευρύ πεδίο δραστηριότητας, καλύπτει την αλληλεία, τις υδατοκαλλιέργειες, τις θαλάσσιες μεταφορές, τον τουρισμό, την αυσιπλοεία, τις κρουαζιέρε. Θα πρέπει κυρίως να στηρίζεται όπως είπαμε στην καινοτομία και στις νέες τεχνολογίες. αυτό σημαίνει στήριξη και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά στήριξη και στην ίδια την ποιότητα. σημαίνει στήριξη στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και σε μορφές τοπικής συνεργασίας. σημαίνει προσπάθεια δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και ανάπτυξης νέων προϊόντων. σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε μια στήριξη της οικονομικής κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην ευρωπαϊκή ένωση. αυτό λοιπόν σημαίνει επιπλέον συνεργασία μεταξύ και των ίδιων των περιφερειών. απαιτείται λοιπόν να υπάρξει ενίσχυση μέσω των διαρθρωτικών ταμείων μέσω του ίδιου του ταμείου της περιφερειακής ανάπτυξης και του ευρωπαϊκού κοινωνικού ταμείου. ευχαριστώ. ευχαριστούμε. παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μιλάμε για τη γαλάζια οικονομία και θα μπορούσαμε να αναφέρουμε πολλά διαφορετικά ζητήματα, γιατί η γαλάζια οικονομία είναι ένας ευρύς τομέας που καλύπτει πάρα πολλά ζητήματα. Προέρχομαι από την Κροατία, μια χώρα που βρέχεται από την Αδριατική και επομένω η γαλάζια οικονομία αντιστοιχεί σε πολύ μεγάλο ποσοστό τη δική μα οικονομία. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να επιμείνουμε στο ζήτημα της ναυπηγίας και θα ήθελα να ρωτήσω τον Επίτροπο Τίμερμανς αν πρόκειται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με εθνικές κυβερνήσεις να χρηματοδοτήσει περισσότερο την Ευρωπαϊκή Ναυπηγία και να καταφέρει να προωθήσει μέσω αυτής την καινοτομία και την απασχόληση. Νομίζω ότι πρέπει να προωθήσουμε την ευρωπαϊκή ναυπηγία. Είναι πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να συνειδητοποιήσουμε ότι πολλές χώρες μπορούν να συμβάλλουν στην ευρωπαϊκή ναυπηγία παράγοντας επιμέρους μέρη πλοίων ή σκαφών. Η ευρωπαϊκή ναυπηγία αντιστοιχεί σε πάρα πολλές θέσεις απασχόλησης και επιθυμούμε να την προωθήσετε. Μάλαγκα για ένα λεπτό παρακαλώ. Eh, ναι, ευχαριστώ πρόεδρε. Επίτροπε για το έργο αυτό το οποίο έχει αναπτυχθεί και είναι ε, πολύ μεγάλη δουλειά σε αυτή την έκθεση με μια επικέντρωση που ε, δίνει μια συνεκτικότητα και πολύ μεγαλύτερη φιλοδοξία και πολλές περισσότερες απαιτήσει. Κάνουμε λόγο για μια ολοκληρωμένη σφαιρική προσέγγιση τώρα που εκινεί από την αηφορία ως κεντρική έννοια και που θέλουμε να αποφύγουμε τους παραδοσιακούς κινδύνους που πολλές φορές ε, ε, ενέχονται στις δράσεις ε, από πλευρά της Επιτροπής. Κάνουμε ρόλο για το, τη δράση και το ρόλο της Ευρώπης που πρέπει να διαδραματιστεί στις θάλασσές μας και στους ωκεανούς. Με συνεκτικότητα, συνάφεια, στρατηγική και συνοχή. Κάνουμε λόγο για την υδατοκαλλιέργεια και την αηφορία Κάνουμε λόγο για τις, ε, την αρχή της πρόληψης στο deep sea mining όσον την ε, εξόριξη ε, μεγάλων, μεγάλου βάθους. Δεν επιτρέπεται να επαναληφθούν τα σφάλματα τα οποία έγιναν στη στεριά. Πρέπει να δείξουμε το σεβασμό μας στη θάλασσα και στον ωκεανό με την καλύτερη στρατηγική για να αντιληφθούμε τις ανάγκες της θάλασσας. Ευχαριστώ. πολύ Πρόεδρε. Ένα από τα προβλήματα σε αυτή τη σύντομη συζήτηση με μικρό χρόνο παρέμβαση είναι ότι δεν μπορεί κανείς να ανταποκριθεί στις υψηλές φιλοδοξίες ε, του θέματος. Ελπίζω ότι μπορούμε να συναγάγουμε τα συμπεράσματα από την αιωλική ενέργεια και να δούμε ποιες νέες τεχνολογίες θα εισαχθούν μετά στη συνέχεια και όχι αντίστροφα. Πρέπει εδώ λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε να δράσουμε σε σχέση με αυτόν τον τομέα και την έρευνα. Ένα άλλο σημείο θα ήθελα να αναφέρω στον χρόνο που έχω την πρόταση για το υγροποιημένο φυσικό αέριο ως ε, μεταβατικό καύσιμο για να βελτιωθεί η κατάσταση του περιβάλλοντος. Ε, ο όρος ε, προσωρινό ή ε, μεταβατικό καύσιμο δείχνει ότι δεν θέλουμε να υπάρξει οποιαδήποτε ολίσθηση όσον αφορά τη δημιουργία ανεργίας. Ευχαριστούμε. σα ευχαριστώ, Πρόεδρε ο σχεδιασμός της οικονομίας και όλοι οι τομείς που συνδέονται με τη θάλασσα και τους ωκεανούς είναι ιδιαίτερα σημαντική υπόθεση. Η κιανή οικονομία δημιουργεί μεγάλο ποσοστό της απασχόλησης εκατομμυρίων ατόμων και έχουμε εδώ και 95 εκατομμύρια ευρώ που συνεισφέρονται η έκθεση σαφώς αναφέρεται στην αλληλοσύνδεση ε, των δραστηριοτήτων στεριάς και θάλασσας, όπου τα στοιχεία αυτά πρέπει να θεωρούνται στοιχεία μιας ε, ενιαίας μεγαλύτερης ενότητας, ενός μεγαλύτερου συνόλου. Και ποιο ε, ποιος είναι ο ρόλος των νέων τεχνολογιών και της καινοτομία στην έρευνα. Ένα άλλο σημείο είναι οι επενδύσεις. Στην έκθεση ασκείται επίκριση ότι ορίζοντας 2020 σε σχέση με τις ε, εξοικονομήσεις ε, ε, πρέπει να καλυφθούν τα κενά και η γαλάζια οικονομία να υποστηριχθεί όπως πρέπει. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Τώρα ο Επίτροπος Τίμερ μας παρακαλώ για να απαντήσει. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή παρότι απουσιάζει και τα μέλη της Επιτροπής Ήτρε για αυτή την ευρεία και πολύ καλοδεχούμενη έκθεση που επίσης αντανακλά τις ε, απόψεις ε, των γνωμοδοτήσεων της Επιτροπής Αλληλείας και Απασχόλησης. Είναι σημαντικό το δυναμικό της ε, κοιανής οικονομίας για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και τονίζεται η σπουδαιότητα των δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης των κρατών μελών για να απελευθερωθεί αυτό το δυναμικό. Η διάσταση της πρέπει πλήρω να εντάσσεται στην προσέγγισή μα. και συμφωνώ απόλυτα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλευρό μου με αυτή την προσέγγιση. Πρέπει να να προστατεύσουμε την ε, διάσταση της αηφορίας ε, στις παράκτιες περιοχές, στις θάλασσες και τους ωκεανούς. Να είναι ε, χωρίς σκουπίδια και χωρίς μόλυνση και ρήπανση οι θάλασσες και οι ωκεανοί. Να μπορεί η έρευνα να αναπτυχθεί, η καινοτομία να αναπτυχθεί. Είναι σημαντικό αυτή η στόχοι να μπορέσουν να υποστηριχθούν με υποστήριξη και των κρατών μελών. Και προαγωγή της καινοτομίας με παραδοσιακές αλλά και καινοτόμες δράσεις και να δούμε τα θέματα της ναυτιλίας και της χαρτογράφησης ε, του πυθμένα της θάλασσας ε, να μπορέσει να προαχθεί η απασχόληση και ε, σε όλο το ευρύτερο πλαίσιο μέσα από τις δράσεις αυτές. Για παράδειγμα, δύο συγκεκριμένα άρθρα υπάρχουν στον κανονισμό του, της του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τις θάλασσες στον ορίζοντα 2020 και το πλαίσιο, πρόγραμμα πλαίσιο για την καινοτομία και την ανάπτυξη. Επίσης το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων δίνει δυνατότητες για προγράμματα και δράσεις σε ε, δράσεις ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου. Ε, μια σωστή αξιολόγηση του εύρους της κιανής οικονομίας πρέπει να γίνει και η αξιολόγηση των δυνατοτήτων. Κάνουμε ήδη τα πρώτα βήματα να διαπιστώσουμε τις διαστάσεις αυτής της κιανής οικονομίας και με τα στοιχεία των στατιστικών υπηρεσιών και οικονομολόγων θα βοηθηθούμε να προχωρήσουμε και να μετρήσουμε και να αξιολογήσουμε την πρόοδο στην προαγωγή των επιχειρήσεων ε, και της ε, δράσης μας επίσης και άλλα στοιχεία όπως ε, να καλύψουμε τα κενά που υπάρχουν όσον αφορά τις δεξιότητες και να μπορέσουμε μέχρι το 2016 να είμαστε αποτελεσματικοί, να δημιουργήσουμε μια πλατφόρμα καινοτομίας ε, για την ναυτιλιακή έρευνα και ανάπτυξη. Συμφωνώ απόλυτα ότι χρειάζεται ένα γενικό πλαίσιο ίσων ευκαιριών και δραστηριοτήτων ώστε να είμαστε πρωτοπόροι στην Ευρώπη Υπάρχει και η εκκίνηση της διαβούλευσης σε ένα ευρύτερο πλαίσιο για αυτά τα οποία πρέπει να πράξει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την αηφόρο χρήση των πόρων στις θάλασσες και τους ωκεανούς και ένα δίκαιο σωστό πλαίσιο το οποίο θα αναπτύξουμε για αυτές τις δράσεις. Ολοκληρώνοντας Πρόεδρε, καλωσορίζουμε ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή την έκθεση. Προσβλέπουμε στο να συνεργαστούμε του σύνεγγυς με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα αυτή τη διάσταση. Ευχαριστούμε. ολοκληρώνοντα τη συζήτηση για την έκθεση αυτή, την οποία θα ψηφίσουμε.